Οι αθεσμικές πραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 69 σε παράγραφος 1 του κανονισμού. Η εκθέσεις που αποτελούν τις εντολές για αυτές τις διαπραγματεύσεις υπάρχουν στο ε, διαδικτυακή σελίδα της Ολομέλειας και οι τίτλοι τους θα δημοσιευθούν στα πρακτικά της Συνόδου. Σύμφωνα με το άρθρο 69 σε παράγραφος 2, ένας αριθμός ε, βουλευτών ή μία οι περισσότερες πολιτικές ομάδες ίσες με το μέσο όρο ε, μπορούν γραπτώς να υποβάλουν μέχρι αύριο το βράδυ τα μεσάνυχτα, 16 Ιανουαρίου δηλαδή, να τεθεί σε ψηφοφορία η απόφαση για έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αν δεν γίνει τέτοιο αίτημα προς την Ολομέλεια, με βά... Ε, όσον αφορά δηλαδή την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ε, μέσα δηλαδή στην προθεσμία που σας ανέφερα, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα μπορεί να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Και τώρα περνάμε